τη ρίζα του προβλήματος σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστούμε την Επίτροπο κύριε Ρέντινγκ. Έξι προτάσεις ψηφισμάτων έχουν κατευθεί και η ψηφοφορία θα γίνει μετά το τέλος ε, των συζητήσεων. Το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης ε, είναι η συζήτηση για την κατάσταση στην Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία. Θα δώσουμε το λόγο ε, στο συντάκτη της γνωμοδότησης. Ένα λεπτό. Συνάδελφος Μιγκάλσκι. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ε, είναι ένα κράτος που έχει αποτύχει. Είναι ένα ε, κράτος ε, στο οποίο δεν μας εκπλήσει που συναντάμε αυτά τα οποία αναφέρονται στο ψήφισμα. Κάνουμε έκκληση να σταματήσουν οι ένοπλες συγκρούσεις, να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι διαπράττουν τα εγκλήματα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ώστε να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση ακολουθούμε μία διτή προσέγγιση, διπλωματική αφενός και αφετέρου από πλευράς της οικονομίας. Είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές, πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ και είναι σημαντικό να το έχουμε κατά νου και γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξουν και παρατυπίες όταν μιλάμε για μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα τα οποία δίνουμε πραγματικά φτάνουν ε, σε αυτούς οι οποίοι τα χρειάζονται. Είναι σημαντική η δυτή προσέγγιση. Ευχαριστούμε κύριε και Συνάδελφος Πρέντα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το θέμα το οποίο συζητούμε αποφασίστηκε την ε, περασμένη εβδομάδα, όπως είναι γνωστό, και τα επακόλουθα θέματα αποφασίστηκαν μόλις τη Δευτέρα, αλλά όταν προτείναμε να έχουμε μία συζήτηση για την ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, υπέρχαν συνάδελφοι που ρωτούσαν, μα είναι επίγον, τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, γιατί θα πρέπει να συζητήσουμε όλο αυτό το θέμα. Όμως όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε διάφορα γεγονότα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και μας έδειξαν ότι βρισκόμαστε σε μια κατεπίγουσα κατάσταση γιατί 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ των υποστηρικτών του πρώην Προέδρου και της, ε, του συνασπισμού της ΕΛΕΚΑ. Και αφού ε, ανέλαβε την εξουσία η ΕΛΕΚΑ, η χώρα βρίσκεται σε χάος, ε, έχουμε καταστροφική κατάσταση και σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά συζητήσαμε και την ε, ε, προειδοποίηση της Βάλερη Άμος. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος Σένισιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία εκτιλήσεται ένα ανθρωπιστικό δράμα, ο συνασπισμός ΕΛΕΚΑ ευθύνεται για ομότητες και βιοπραγίες. 70% του άμαχου πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας και αναγκάζεται να διαφεύγει στη σαβάνα και στη ζούγκλα. Υπάρχουν πάρα πολλές αρρώστιες και πρέπει να διασφαλίσουμε ό,τι, ό,τι λέγω ότι θα μπορέσουμε να προηθμηθεύσουμε τουλάχιστον ιατρική βοήθεια σε αυτόν τον πληθυσμό αλλά και πολιτική υποστήριξη και γενικά ανθρωπιστική βοήθεια. ιδιαίτερα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης με στόχο να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός έτσι ώστε να μπορέσουν να οργανωθούν ελεύθερες εκλογές η συλλογή παρανόμων όπλων ο αφοπλισμό μάλλον είναι κάτι που επίση πρέπει να υποστηρίξουμε. Ευχαριστούμε κυρία Συνήση, τώρα κυρία Όγιολάντ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πέρασαν σχεδόν έξι μήνες από τότε που έγινε η το αντισυνταγματικό πραξικόπημα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Η Ένωση επανειλημμένω έχει εκφράσει την ανησυχία τη για την απουσία κράτου δικαίου και για την ανάγκη να επανέλθει η ασφάλεια στον άμαχο πληθυσμό. Το δικαστικό σύστημα πρέπει να μπορέσει να τιμωρήσει όσους έχουν παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλαίως θα χρειαστεί διεθνής παρέμβαση όπως είπε περασμένο μήνα και το Διεθνές Δικαστήριο και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία πρέπει να τύχει αποστρατιωτικοποίησης τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Όγιολαντ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Βερζιά. Ε, είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από την 11η Ιανουαρίου που έγινε το πραξικόπημα και ανέλαβε ο Μισελο ο αρχηγός των ανταρτών της ΕΛΕΚΑ, τι βλέπουμε, ότι σήμερα ο βασιλεύς είναι γυμνός, γιατί φαίνεται ότι δεν ελέγχει τίποτα η ΣΕΛΕΚΑ, όπως δείχνουν οι πρόσφατες βιοπραγίες. Η Γαλλία που έχει τσαδικό παρελθόν έχει ιδιαίτερη ευθύνη. Αρνείται όμως να παρέμβει. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα για τη σημαντική βοήθεια που χορήγησε η Ένωση στη χώρα αυτή η ανθρωπιστική κατάσταση θα χειροτερέψει. Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται άμεση βοήθεια. Ενώ η βοήθεια δεν φτάνει μόνο, παρά μόνο στο 20% της περιφέρειας της χώρας. Δεν ξέρουμε πια ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Ευχαριστούμε κυρία Βεριά. Συνάδελφος Λόχμπίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι πολίτες στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία υποφέρει. Υποφέρει μετά από χρόνια αγώνων μεταξύ οπλισμένων ομάδων, ενόπλων ομάδων ε, και του στρατού. Το 2012 ε, πολλές ενόπλες ομάδες είχαν δηλώσει ότι ε, τελειώνουν, τελειώνουν οι εχθροπραξίες. Παρ' όλα αυτά συνεχίζονται οι σειράξει, Έχουμε εξοδικαστικές ε, εξοδικαστικές εκτελέσεις, ε, βιασμούς ε, γυναικών και βασανιστήρια και κακοποίηση. Πολλέ πολλές ένοπλες ομάδες στρατολογούν παιδιά για να πολεμούν στο πλευρό τους. Οι αριθμοί μας ανησυχούν ιδιαίτερα και αποδεικνύουν ότι οι έθραυστες δομές του νόμου και της τάξης έχουν καταρρεύσει. Δεν υπάρχει σύστημα δικαιοσύνης. Επί πολλά χρόνια υπάρχουν βίες σειράξεις και δεν ε, λειτουργεί σχεδόν ουδόλως η κυβέρνηση πολλοί πολίτες έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους και την πατρίδα τους για να μπορέσουν να ζήσουν. 1,6 εκατομμύρια πολίτε ε, διατρέχουν κινδύνο και δεν μπορούν ε, να έχουν τα απαραίτητα για τη διατροφή τους, ε, δεν έχουν ούτε καν νερό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να υποστηρίζει με ανθρωπιστική βοήθεια και να προσπαθήσει να βελτιώσει την κατάσταση ώστε η κυβέρνηση να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα να συλλητεύσουμε τις περιπτώσεις παραδείας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι διατάσσουν και αυτοί οι οποίοι διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει αυτούς που υπεραμείνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Λόχ Μπίλερ. Ε, οι συντάκτες ε, έλαβαν το λόγο και δίνουμε τώρα τους, στους συναδέλφους εκ μέρους των ομάδων το λόγο. Η συνάδελφος Γκάμπριελ τον Ιούνιο χαιρετήσαμε τα δείγματα βελτίωση στο πολιτικό επίπεδο για την Κεντροφυρκανική δημοκρατία, αλλά υπογραμμίσαμε ότι η κατάσταση ό,τι αφορά την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ εύθραστη και πάλι είχαμε δίκιο. Δυστυχώ σήμερα η διαδικασία οικοδόμηση και θεστεροποίηση τη χώρα αμφισβητείται. Εκτίθενται κάποιε προτεραιότητε, η ανθρωπιστική κρίση, θίγει πλήττει 1,6 εκατομμύρια άτομα και θα πρέπει να προσφέρουμε και πάλι υπηρεσίες σε βάση. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των παιδιών στρατιωτών. Υπάρχει και η στρατιωτική πτυχή που είναι πρωταρχική. Θα πρέπει να γίνει συλλογή όπλων ορθά σε, όλες τις, σε όλη τη χώρα. Επίσης, οι συμφωνίες της Λίμπρεβιλ παραμένουν σημείο αναφορά. Εμεί απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους εταίρους διεθνεί και περιφερειακούς να ενισχύσουν τη δράση του ε, για να ενισχυθεί η κοινή δράση. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Γκαμπριέλ. συνάδελφο. Ρεπό. Είναι δεύτερη φορά που φέτος το Κοινοβούλιο συζητάει την κατάσταση στα ανθρώπινα δικαιώματα στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Εδώ και δεκαετίες η χώρα αυτή ήταν από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου και πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι από τις κυριότερες αξίες της Ένωσης αλλά και της Συμφωνίας Κοτονού. Η Ένωση κρατάει στα χέρια της ένα σημαντικό εργαλείο μέσω της σύμβασης αυτής και βλέπουμε ότι η αστάθεια στη χώρα αυτή που αναγκάζει τον κόσμο να φεύγει από τα σπίτια του και σημειώνονται συνεχώς όλο και περισσότεροι βιασμοί έχει καταστήσει τα πράγματα αφόρητα πρέπει η Ένωση να υποστηρίξει πλήρως την απόφαση να ερευνηθεί η κατάσταση εκεί είναι σημαντικό και για τα θύματα και τις οικογένειές τους τα εγκλήματα αυτά να τύχουν μια σωστή έρευνα και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Όμπερμα τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τότε που απέσπασαν την εξουσία τα μέλη της, του συνασπισμού ΣΕΛΕΚΑ έχουν διαπράξει πάρα πολλά εγκλήματα και έχουν αυθαίρετα στρατολογήσει πολίτες σε όλες τις επαρχίες. Αυτός ο συνασπισμός σε ΛΕΚΑ θα πρέπει να καταδικαστεί από την διεθνή κοινότητα και θα πρέπει να καταδικαστούν τα εγκλήματα πολέμου θα πρέπει να δικαστούν σύμφωνα με το εθνικό αλλά και σύμφωνα με το διεθνές ποινικό δίκαιο. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ασχολείται ήδη με την κατάσταση στην Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία και θα πρέπει και τα εγκλήματα πολέμου να στυλιτευθούν. Δεν θα πρέπει να υπάρξει παραγραφή για τα δικήματα κατά των, της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Όμπερ Μάγερ. Εκ μέρου ε, των ομάδων ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις. Οι υπόλοιποι βουλευτέ τώρα ο συνάδελφο Κέλλη. Ε, Συζητούμε τώρα το θέμα της κεντροφερκανικής δημοκρατίας εδώ σήμερα ε, με μεγάλη ανησυχία και αυτό κυρίως επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυρίως δωρητής για τη χώρα αυτή δίνει πάνω από 20 εκατομμύρια το χρόνο αν και η δημοκρατία κέρδισε την ανεξαρτησία της ε, πριν αρκετό καιρό, ποτέ στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ειρήνη στη χώρα. σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους η χώρα αυτή είναι πάρα πολύ πλούσια. Όμως ε, γι' αυτό και ακριβώς το λόγο δεν είναι κατανοητό γιατί είναι τόσο μεγάλη η φτώχεια στη χώρα. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να τεθεί τέλος στη βία. Πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά για να σημειωθεί πρόοδος στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κέλλη, συνάδελφος Ευχαριστώ η κεντροαφρικανική δημοκρατία έχει βυθιστεί στο χάος και αυτό έχει οδηγήσει σε συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως από τότε που ανέλαβαν την εξουσία ε, οι αντάρτες της ΕΛΕΚΑ. Αυτοί ουσιαστικά λατούν τη χώρα προβαίνουν σε και σε κτηνοδίες. Είδαμε ανθρώπους ε, να πεθαίνουν από την πείνα και υπάρχει διάλυση σε ολόκληρη τη χώρα παρόμοια με αυτό που είδαμε στη Σομαλία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τώρα διεθνή στρατιωτική επέμβαση για να έχουμε ειρήνη στη χώρα και να σταματήσουν οι οι οπαδοί της Τζιχάντε να έρχονται από το βορρά. Ως προτεραιότητα πρέπει να παγιώσουμε την εντολή που έχει δοθεί στις διεθνείς ειρευνητικές αποστολές και πρέπει να παράσχουμε και αρρωγή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ευχαριστούμε την κυρία Κρατήρια και την κυρία Μακοβέη. Sunt foarte îngrijorată πάρα πολύ για την κατάσταση του πολέμου και της ατιμορρησίας που φαίνεται να κυριαρχεί στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Φαίνεται άνθρωποι να πεθαίνουν, να βασανίζονται για κανείς δεν αντιδρά. Η διεθνής ε, κοινότητα παρακολουθεί σιωπηλά αυτή τη νέα κρίση στη χώρα. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη εσωτερική σύραξη, έχουμε 240.000 πρόσφυγες και έχουμε και 100.000 παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση ή έχουν αναγκαστεί να γίνουν στρατιώτες. Ε, έχουν ξεκινήσει τώρα έρευνες ε, για το τι συμβαίνει στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αλλά το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ισχύει για όλες τις χώρες, ακόμη και για τις χώρες που έχουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο λαό της Κεντροφρικανικής Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένουμε ποιο θα βγει νικητής από τη σύραξη και να υποστηρίξουμε τελικά όποιον νικήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μακοβέη και περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω περισσότερους ε, συναδέλφους που ζητούν το λόγο από όσους μπορούν να μιλήσουν τελικά. Σας ζητώ την κατανόησή σας λοιπόν, συνάδελφος ε, Λίτσεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η κατάσταση στην Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και φαίνεται ότι χάνουμε τον έλεγχο. Οι συγκρούσεις ε, μεταξύ, τους, ε, μεταξύ των εκπροσώπων του πρώην Προέδρου Πασίζη και των ε, τωρινών έχοντων την εξουσία εντείνονται. Είναι χιλιάδες τα θύματα και από την δύναμη ΦΟΜΑΚ, από την πολυεθνική δύναμη της Κεντρικής Αφρικής. Θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να αναλάβει δράση για να τεθεί ένα τέλος σε αυτή τη σύγκρουση. Ευχαριστούμε κύριε Λίσεκ. Συνάδελφος Γκέριγκερ Ντεόντεμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε εφόσον από τότε μάλλον που άρχισε, ανέλαβε την εξουσία ο συνασπισμός ΕΛΕΚΑ, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η βία, οι βιασμοί και οι λαιλασίες ε, έγιναν σύνηθες φαινόμενο. Πράγμα που οδήγησε σε αποχώρηση, έξοδο των του πληθυσμού πολλών περιφερειών και εγκαταλείφθηκε η γεωργία και η λειτουργία του κράτους βέβαια καθώς και οι ιατρικές υπηρεσίες. Ένα τρίτο του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί, μετατοπιστεί και χρειάζεται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. 100.000 χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια, η ανέχεια είναι τρομερή, τα παιδιά υποφέρουν ιδιαίτερα και έχουν αναγκαστεί πολλά από αυτά να μπουν στο στρατό η διεθνής κοινότητα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη παρουσία εκεί. Ευχαριστούμε την συνάδελφο Γκέριγκερ Ότεμπερκ. Η συνάδελφο Εσαγιά κλείνουμε τη διαδικασία κατσουδιάη. Ευχαριστώ. Η κυβέρνηση στην Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία έχει σχεδόν καταστραφεί και είναι πάρα πολύ ανησυχητική η κατάσταση. Εκτός της πρωτεύουσα ε, δεν υπάρχει αστυνομία, ε, δεν, υπάρχει δεν υπάρχουν δικαστές ε, και η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει από τις πόλεις και τα χωριά και τρώνε ρίζες. Τους πλήττει ελονοσία, γυναίκες πεθαίνουν στη γέννα και η πείνα σκοτώνει τους ανθρώπους περισσότερο από τον πόλεμο, από την σύγκρουση. Είναι πραγματικά τρομακτικό ότι η ότι κοινότητα φαίνεται να μην δείχνει καμία προσοχή για το τι συμβαίνει στη χώρα και όπως είπαν καλοί συνάδελφοι προηγουμένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως δωρητή ε, δεν μπορεί να αποποιηθεί των ευθυνών τη. Χρειαζόμαστε κατεπήγοντα μέτρα για να σώσουμε ανθρώπινε ζωέ στη χώρα. Ευχαριστούμε τη συνάδελφα εσαγιά, Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch και τώρα θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ. Πρόεδρε, η Επιτροπή χαιρετίζει το σχέδιο ψηφίσματος, διότι η κατάσταση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική από την έναρξη της κρίσης το Δεκέμβριο του 2012 πάνω από πέντε μήνες ε, μετά την ε, μη συνταγματική αλλαγή κυβέρνησης ε, και τώρα η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κινείται προς μια κατάσταση αναρχίας. Μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο σκοτώθηκαν πάνω από 60 άτομα στην βορειοδυτική χώρα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κλιμάκωση της βίας. Καταδικάζουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συνεχίσουμε μέσω κάθε δυνατού διάβλου να καταπολεμούμε την ατιμορρησία. Αυτό θα το κάνουμε μαζί με τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους μας και με τα διεθνή βήματα όπως είναι ναι, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Η Αντιπρόεδρος ε, κυρία Άστον έχει ε, ε, εκφράσει τη λύπη της το Μάρτιο του 2013 με μια δήλωση και λέει ότι είναι πεπισμένη ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι διαπράττουν τα εγκλήματα. Ζητάμε από τις μεταβατικές αρχές στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να αποκαταστήσουν τον νόμο και την τάξη, να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό και να είναι συμβατή με τη συμφωνία της Λιμπροβίλ. Επίσης υποστηρίζουμε τη δημιουργία ε, της ε, ε, ειρηνευτικής προσπάθειας που γίνεται υπό την αιγίδα της Κεντρικής Αφρικής και υπέρ του προγράμματος σταθεροποίησης που χρηματοδοτείται από το μέσο σταθερότητας. Παρά την, το τεράστιο μέγεθος της τωρινής κρίσης, η κεντροαφρικανική δημοκρατία διατρέχει τον κίνδυνο να ξεχαστεί ως περιοχή κρίσης, αλλά δεν θα ξεχαστεί και χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ξεχαστεί. Θα υπάρξει κινητοποίηση διεθνώς, ούτως ώστε η κεντροαφρικανική δημοκρατία ε, να τεθεί ως προτεραιότητα και θα συζητηθεί και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών με αυτή την προτεραιότητα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω μια δήλωση της 10 Σεπτεμβρίου της συναδέλφου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα που καταδικάζει τη δολοφονία ε, της Act και της ανθρωπιστικής οργάνωσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απολύτως απαράδεκτο το να γίνονται στόχοι άνθρωποι που προσπαθούν να σώσουν τις ζωές άλλων ανθρώπων και έχουμε εκφράζουμε τη συμπαθιά μας προς τις οικογένειες ε, των θυμάτων. Θα πρέπει να είναι βασική αρχή μας το να τηρούνται οι ανθρωπιστικέ αρχέ. Το θέμα της ασφάλειας έχει γίνει κέριο πρόβλημα. Περιορίζει τη δυνατότητα των εργαζομένων ε, στον τομέα τη επιστημικής και ανθρωπιστικής βοήθειας ε, να μετακινηθούν. Οι, εκτελέσει, ε, η σωματική βία συμπεριλαμβανομένη τη σεξουαλική βίας, οι εκβιασμοί, η παράνομη φορολογία, λασίε, αρπαγές επηρεάζουν τη ζωή της χώρας ολόκληρης και ένας πληθυσμός που ήδη βρίσκεται στα όρια της φτώχειας ε, οθείται στα όρια του. Η Επίτροπος Γεωργίευα οργανώνει μια συνάντηση υψηλού επίπεδου σε υπουργικό επίπεδο ε, στις 25 Σεπτεμβρίου για να ε, ευαισθητοποιηθούν όλοι για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να βοηθά με το στενό συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους ώστε να καταλήξουμε σε σταθεροποίηση της χώρας και σε υποστήριξη της πολιτικής διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επίτροπο Ρέντινγκ. Ολοκληρώνει τη συζήτηση για το ψήφισμα αυτό. Έξι προτάσεις ψηφίσματος έχουν κατατεθεί και η ψηφοφορία θα γίνει μετά την συζήτηση των ψηφισμάτων. Το επόμενο σημείο είναι το ψήφισμα